Κοινοβουλίου στο πώς επικεντρώνει την προσοχή του στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων από όλους τους εταίρους. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ψηφίσουμε για τις προτάσεις ψηφισμάτων, αφού ολοκληρώσαμε τη συζήτηση. Ψηφίσουμε καταρχάς το ψήφισμα για την Νότια Αφρική σφαγή απεργών ανθρακορίχων. Έχουμε όμως έτοιμα επί της διαδικασίας. Κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν επιτρέψατε γιατί δεν δώσατε τη δυνατότητα ε, να λάβουμε το λόγο στη συζήτηση. Δεν πρέπει να ακολουθούμε μια δημοκρατική διαδικασία. Εγώ στράφηκα ε, στο συνεργάτη σας ζητώντας τη διαδικασία Catch the να μιλήσω και εσείς με αγνοήσατε πλήρω. Θέλω να μου εξηγήσετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος. Δεν είχα δει ότι το όνομά σας είναι. Μάλλον είχα δει, αλλά δεν μπορούσαμε να δώσουμε σε πάνω από δύο άτομα. So the and Είχαν κάποιοι ε, ζητήσει το λόγο πριν από εσά και δεν μπορούσα να σα δώσω και εσά το λόγο. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην εξέταση πρόταση ψηφίσματο από έξι πολιτικέ ομάδε. Δεν υπάρχουν τροπολογίε. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματο. Ψηφί υπέρ. Again. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενο θέμα είναι η ψηφοφορία προτάσεων ψηφίσματος για τη δίωξη των μουσουλμάνων Ροίγκια στη Βυρμανία. Θα ψηφίσουν καταρχάς το κοινό ψήφισμα από έξι πολιτικές ομάδες. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Θέτω το κοινό ψήφισμα σε ψηφοφορία. Ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενο θέμα είναι η ψηφοφορία επί προτάσεων ψηφίσματος για το Αζερμπαϊτζάν, την περίπτωση του Ραμίλ Ζαφάρου. Ψηφίζουμε καταρχάς κοινό ψήφισμα από πέντε πολιτικές ομάδες. Και εδώ έχουμε τροπολογίες. Τροπολογία 1. Ονομαστικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 των πρασίνων Ονομαστικά ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία. Τροπολογία 4. Ονομαστικά και αυτή η του ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Τροπολογία 7 γίνεται δεκτή. Τροπολογία 8 ψηφίζουμε ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η τροπολογία 8. Ψηφίζουμε την τροπολογία 6 και την αναθεωρημένη 12 που είναι ταυτόσιμες ε, ψηφίζουμε ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 11 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τροπολογία 13 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. τροπολογία εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ψηφίζουμε ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Η τροπολογία ναι, έχει αποσυρθεί. Και τώρα ψηφίζουμε το, την κοινή πρόταση ψηφίσματος συνολικά με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τα πρακτικά της συνεδρίασης θα υποβληθούν ε, ε, στο Κοινοβούλιο για έγκριση. Αν δεν υπάρχουν ε, ενστάσεις, ε, οι προτάσεις ψηφίσματος που εγκρίθηκαν σήμερα θα διαβαστούν αρμοδίως. Και εδώ μπορώ να κηρύξω τη λήξη των εργασιών της Ολομέλης αυτής.